Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, κυρίως στην έναξη της σημερινής συνεδρίασης και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα μια ε, αντιπροσωπεία από τα 16 κρατήδια εκπρόσωποι των Πρασίνων ε, αρμόδιοι για θέματα μεταφορών. Δύο φορές το χρόνο συνεδριάζουν και αυτή τη φορά έχουν έρθει στις Βρυξέλλες. Ε, καλώς ορίσατε, είναι της, ε, του κόμματος των Πρασίνων και της Συμμαχίας των 90. Και μετά από αυτή την καταπληκτική εισαγωγή περνούμε στη μερίσια διάταξη. Πρώτον, έγκριση της προσωνής ημερήσιας διάταξης μπορεί να εγκριθεί ε, αν δεν έχει κάνει καμία αντίρρηση, οπότε βλέπω όχι, οπότε εγκρίνεται και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσει, μπορούν να θεωρηθούν εγκεκριμένα και τα πρακτικά τη 14ης, 15 η Μαρτίου και τη 7 η Απριλίου 2016. Ανακοινώσει του Προέδρου Προ το παρόν δεν έχω και περνούμε αμέσως στο σημείο 4 πρόταση για κανονισμό για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια ε, στη θάλασσα. Η, ε, η συγκίτρια είναι η κυρία Μαρίν Κριστίν Αγνοτού, η οποία έχει αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, συνάδελφοι, αν διαβάσει κανείς τα πρακτικά της συνάντησης του Συμβουλίου Υπουργών της 21ης Απριλίου, ε, δεν χρειάζεται να σας παρουσιάσω τίποτα γιατί από ό,τι φαίνεται όλα έχουν προαποφασιστεί. Θα πρέπει να τεθεί ένα ερώτημα όμως εδώ. Ποιος αποφασίζει εμείς που εκπροσωπούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της χώρας μας ή μήπως είμαστε όλοι υπό τις διαταγές του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ο κύριος Αβραμόπουλος, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είπε ότι εμπιστεύομαι την δυνατότητα ολοκλήρωσης της νομοθετικής διαδικασίας για τη δημιουργία ενός νέου ε, συνοριοφυλακού σώματος πριν από τον Ιούνιο. Το κείμενο το οποίο υιοθετήθηκε ε, τίνει να διαβεβαιώσει αυτούς οι οποίοι ε, στη δική μου πολιτική ομάδα σαν παράδειγμα θεωρούν ότι οι αρχές της εθνικής κυριαρχίας θα τεθούν σε αμφισβήτηση γιατί το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο και όχι από την Επιτροπή. Στο Συμβούλιο εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη. Λέγεται στην απόφαση ότι θα πρέπει να αποφύγουμε ένα χάος στα εξωτερικά σύνορα που θα οδηγήσει στο τέλος της ελεύθερης διακίνησης στα πλαίσια του χώρου Σέγγεν. Βασική ανησυχία δεν είναι λοιπόν η προστασία των σύνορων των κρατών μελών, ούτε όπως θα θέλατε πολλοί από εσά η προστασία των μεταναστών, ένα επιχείρημα το οποίο είναι ο λίγων μη ειλικρινές σε επίπεδο διανοητικό γιατί δείχνει ότι ζούμε σε ένα κόσμο εκτός πραγματικότητας. Γιατί ακόμα και αν εμείνουμε σε αυστηρά οικονομικά κριτήρια, καμία από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σε θέση να υποδεχθεί ε, βήμ, ε, κύματα μεταναστών όπως προβλέπουν οι υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών. Συνεπώς λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μια σωστή λύση, βλέπουμε την φτώχεια όμως των ε, συμπατριωτών μας, η οποία αυξάνεται συνεχώς. Φυσικά πρέπει να έχουμε και καρδιά όταν ασκούμε πολιτική, αλλά πρέπει όμως να είμαστε υπεύθυνοι στις αποφάσεις που παίρνουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Πολλοί από εσά με κατηγόρησαν ότι δεν διαφοροποιώ τους παράνομους μετανάστες από τους νόμιμους μετανάστες. Εδώ θα πω τα στοιχεία του Frontex. Το 2015 υπήρξαν 1.083.000 παράνομες είσοδοι στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η τεράστια πλειοψηφία στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Σύμφωνα με τους αριθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 17 άλλα 3 εκατομμύρια. Η υπηρεσία Frontex λέει ότι το Μαρόκο που παράγει φυσικά κάναβη είναι η πρώτη χώρα από τις οποίες προέρχονται οι εκμεταλλευτές και μεταφορείς παράνομων μεταναστών. 32.000 Μαροκινοί ζουν στην Ευρώπη ε, σε επίπεδο χωρίς κάλυψη, νόμιμη θα έλεγα και αυτό κάτι δείχνει. Ε, οι προϋπολογισμοί τώρα για την προστασία των συνόρων στην Αυστραλία για 26.000 χιλιόμετρα θαλάσσια σύνορα. Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται είναι 4,7 δις το χρόνο με 8.000 υπαλλήλους. 5.000 παράνομοι είσοδοι, ε, σήμερα 100.000 ε, ε, πριν εφαρμοστεί η νέα πολιτική που λέγεται No Way. Στις Ηνωμένε Πολιτείες για 20.000 χιλιόμετρα επίγειων συνόρων. Η Υπηρεσία Προστασίας των Συνόρων έχει προϋπολογισμό 12,5 δις το χρόνο με 36.000 υπαλλήλους. 400.000 παράνομοι μπαίνουν το χρόνο στις Ηνωμένε Πολιτείε και αυξήθηκε όταν ο πρόεδρος Ομπάμα το 12 έδωσε χαρτιά σε πάρα πολύ κόσμο και από εκεί και πέρα βέβαια δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα όπως και μετά από αυτό που έκανε η Μέρκελ στη Γερμανία. Αν συγκρίνουμε λοιπόν την κατάσταση, θα δούμε ότι στο Σέγγεν για 42.000 χιλιόμετρα θαλάσσια έχουμε 115 εκατομμύρια προϋπολογισμό του Frontex με 400 που θα φτάσει τα 330 και θα οδηγηθούμε σε 1.000 μονίμους υπαλλήλου και 1.500 τους οποίους θα παρέχουν τα κράτη-μέλη για τη δύναμη τοχείας παρέμβασης. Ένα εκατομμύριο 800.000 ήταν οι παράνομοι που μπήκαν στην Ευρώπη τον προηγούμενο χρόνο. Κοιτάξτε μόνο οι αριθμοί. Λένε ότι αυτή η νέα υπηρεσία δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει μια σωστή και φιλόδοξη πολιτική διαχείριση των συνόρων μας. Για να έλθω σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπαραντίκα, η οποία αντέγραψε αυτά που είπε ο κύριος Τίμερμανς αλλά νομίζω ότι δεν είναι παρά κάτι το οποίο ε, θα παραμεριστεί από μόνο του όταν η κρίση διευρυνθεί. Η έκθεσή μου δεν είναι μια επίθεση εναντίον των μεταναστών και λυπάμαι γιατί πολλοί από αυτούς ε, αδιαφορούν όταν διαβάζουν τη συνέντευξη του κ. Μακδόναλντ της Europol, ο οποίος λέει ότι 10.000 ανήλικοι μετανάστες έχουν εξαφανιστεί και τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης σε δίκτυα πορνείας. Εσείς θέλετε να συνεχίσετε λοιπόν να τροφοδοτείτε αυτήν την απαράδεκτη πολιτική για τη μετανάστευση, την ασυνείδητη πολιτική ή μήπως να εγκαταλείψετε τις ιδεολογίες και να σκεφτείτε το μέλλον της χώρας σας, των παιδιών σας και των πολιτών σας. Γιατί θέλετε να γίνει δεκτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ μας οδηγεί σε κατευθύνσεις τις οποίες εγώ κρίνω ιδιαιτέρως επικίνδυνες γιατί μας απομακρύνει ακόμα περισσότερο από την εθνική μας κυριαρχία. Μήπως χρειάζεται να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Μήπως χρειάζεται να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας. Οι χώρες μας απειλούνται, απειλούνται όλες. Ας εγκαταλείψουμε λοιπόν τα ωραία αισθήματα και ας μην μείνουμε στο Frontex, αλλά ας εκμεταλλευτούμε τα στοιχεία του Frontex που είπε ότι έγινε αντικείμενο χρήσης και κατάχρησης από το ISIS η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η έκθεση του 16. και ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας της Ομοσπονδιακής Γερμανίας λέγει σε μια συνέντευξή του ότι οι γερμανικές υπηρεσίες έκαναν λάθος όταν δεν θεώρησαν ότι θα χρησιμοποιούσαν τα κύματα των μεταναστών ή του ISIS και ότι η Γερμανία σήμερα αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο τρομοκρατικό κίνδυνο στην ιστορία της. Ο χώρος Σέγγεν μας εκθέτει σε πολύ περισσότερους κινδύνους από ό,τι σε ωφέλη. Il a été dit euh, εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε χρυσά κλειδιά για να σώσουμε τον κόσμο, αλλά χάσαμε το πρόχειρο μικρό κλειδί για να λύσουμε το δικό μας πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με την κρίση αυτή να αναλάβουμε τις ευθύνες μας πριν να ασχοληθούμε με το να διορθώσουμε τα κακά του κόσμου γύρω μας. Λοιπόν, αυτό σαν στόχος δεν είναι κακό, αλλά οι λύσεις τις οποίες προτείνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν είναι στο ύψος της χρυσή κλίδας των περιστάσεων. Θα τελειώσω απευθυνομένη κυρίως στους Γάλλους συναδέλφους, αν και δεν βλέπω και πολλούς στην αίθουσα, και ιδιαίτερα αυτούς που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στους Ρεπιμπλικές στη Γαλλία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε διπλή γλώσσα. Πολλοί από αυτούς εκφράζουν διαφορετικές γνώσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτές που εκφράζουν στις εκλογικέ του περιφέρειες στη Γαλλία. Θα είμαι λοιπόν πολύ προσεκτική σε σχέση με την εκλογική του συμπεριφορά για την έκθεση που ακολουθεί. Πρέπει να σεβαστούμε τη δημοκρατία, πρέπει να σεβαστούμε την εθνική κυριαρχία των χωρών μας. Αυτό θα διατηρήσει την Ήπειρο στην Ευρώπη, αυτό θα φέρει την ευμάρεια στους Γάλλους πολίτες και φυσικά και στους υπόλοιπους πολίτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο κυρία Νοτού για το σχέδιο έκθεσής της Για το περιβάλλον, ε, ε, περιεχόμενο συγγνώμη και το ύφο θα πω δύο πράγματα στη συνέχεια. Πάντως είναι καλό, πιστεύω, να καθίσουμε να καταλάβουμε ότι η τραγωδία των ετούντων άσυλο, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, τις τελευταίες εβδομάδες αυξάνεται συνεχώς, τεράστια αύξηση. Η συμφωνία με την Τουρκία μοιάζει να λειτουργεί, ας το πούμε έτσι, αλλά ο αριθμός σκαφών που φεύγουν τώρα από τη Λιβύη και άλλες χώρες τη Βορείου Αφρικής προς την Ιταλία, τη Μάλτα, τη Λαμπεντούζα, αυξάνεται ραγδαία με όλα τα συμπαραμαρτούντα ε, ρίσκα. Μπορεί να λέει η κυρία Αρνοτού ότι δεν στρέφεται κατά των μεταναστών, αλλά όταν την ακούει κανείς και διαβάζει και την έκθεση, τότε ε, πραγματικά ε, βάζει όλους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στο ίδιο τσουβάλι. Χρειάζεται εδώ τεράστια προσοχή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολιτικοί ε, πρόσφυγες, που διώκονται και ζητούν άσυλο. Υπάρχουν οικονομικοί πρόσφυγες και βεβαίως υπάρχουν και εγκληματικά στοιχεία και ενδεχομένως και τρομοκράτες μεταξύ αυτών. Αλλά τώρα να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Πραγματικά εμείς έχουμε πρόβλημα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως ομάδα. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Μετά, έρχομαι τώρα στην ουσία της έκθεσης. Κοιτάξτε, η Επιτροπή Ελευθεριών αλλά και η δική μας Επιτροπή Μεταφορών βιάζονται να ε, περάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η αναθεώρηση του κανονισμού έτσι ώστε ε, ο οργανισμός να μπορέσει σωστά να ανταποκρίνεται στο έργο του και να σώνει ζει και ανθρώπους. Αυτά που ζητάει η κυρία Ορνοτού αποδυναμώνουν όλο και περισσότερο ε, την ευρωπαϊκή συνεργασία. Δεν ομιλεί η συγγήτρια για κοινοτική συνεργασία, ε, αλλά για διακρατική, διακυβερνητική. Λέει τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν το α, το β και τα λοιπά. Αυτό είναι εις βάρος του κανονισμού. Για το Σέγγεν τώρα δύο λόγια. Ε, στην αιτιολογική έκθεση λέει η κυρία Αρνονότου ότι ήταν μια επιπολαιότητα το Σέγγεν, εν πάση περιπτώσει κάτι που δεν το κάναμε μετά από όρημη σκέψη και θα πρέπει επιγόντω αυτά τα πράγματα να επιστρέψουν στα χέρια των κρατών μελών. Εμεί το ΕΛΚ δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα δεχτούμε αυτά. Το ΕΛΚ τι λέει, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και των θαλασσίων ε, στη νότια όχθη μας. Αλλά στο εσωτερικό της Ευρώπης όσο γίνεται θα πρέπει να είναι ανοιχτά τα εσωτερικά σύνορα. Αυτό είναι κατάκτηση και κεκτημένο και έχει και τεράστια οικονομική σημασία εκτό των άλλων. Τέλο, Πρόεδρε, να πούμε και δύο λόγια για τον προπολογισμό. Νομίζω ότι η κυρία Νοτού εδώ έχει κάποιο δίκιο ότι ο προπολογισμό και τη Frontex και του ΕΜΣΑ αλλά και του Οργανισμού για την Αλία υφίσταται τεράστια πίεση. Ιδιαίτερα αν το συγκρίνεται πούμε, με υπολογισμού που έχει η Αυστραλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω να απαντήσει σε σχέση με αυτό, πώς σκέφτεται να τα εφαρμόσει στην πράξη. Συμπέρασμα και συνοψίζοντας. Το ΕΛΚ είναι υπέρ της ενίσχυσης ε, του οργανισμού ΕΜΣΑ, αλλά δεν μας αρέσει το ύφος ε, της έκθεσης της συναδέλφου μας από την ΙΕΝΕΦ. Αυτό είναι και στην γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΛΥΒΕ. Δεν είναι το ύφος κάτι που μας καλύπτει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λούση Άντερσεν. Γιατί δεν είναι παρόν ο κ. Φλέκενστάιν από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Μάλιστα, ναι, ομιλώ εκ μέρου του Φλέκενστάιν. Σε ό,τι αφορά την έκθεση, θεωρούμε ότι το σχέδιο και η, ε, ε, η, συγκεκριτική έκθεση είναι πραγματικά ε, ιδιαίτερα επιθετικού χαρακτήρα. Αυτά μάλιστα απλά μετά από μια σύντομη ανάγνωση του, της εισηγητικής εκθέσεως, η οποία στιγματίζει τους ε, ε, μετανάστες. Και μάλιστα αυτό διαχέεται και σε όλο το κείμενο. Θεωρούμε μάλιστα ότι η έκθεση ξεπερνά κατά πολύ τις, ε, τα όρια των αρμοδιοτήτων της εισηγήτριας. Ορισμένα μάλιστα είναι και νομικώς προβληματικά, ιδίως όταν μιλεί για τύπου τροπολογιών που προτείνει, δηλαδή για συμπερίληψη πραγμάτων που κανονικά θα έμπαιναν σε κανονισμό, για παράδειγμα για επικοινωνιακέ εκστρατείε. Πάντω, οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε αποφάσισαν να μην ασχοληθούν διόλου με την εισηγήτρια και να καταψηφίσουν το σχέδιό τη στο σύνολό του. Στην ε, ουσία στηρίζουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρούμε ότι έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα και στοχεύει όντω να στήσει τα πόδια της μια ενισχυμένη συνεργασία, όπως άλλωστε είπε και ο συνάδελφός μου του Λαϊκού Κόμματος. Νομίζουμε ότι συμβαδίζει άλλωστε και με τις προτάσεις του, των ε, οργάνων που φυλάσσουν τα σύνορα, καθώς και ε, των αρχών για την Αλία. Έχουμε και γνωμοδότηση για την ε, ακτοφυλακή στην Επιτροπή Θεμελιωτών Ελευθεριών για συνεργασία που νομίζουμε ότι η ΕΜΣΑ μπορεί όντω να υλοποιήσει με ρεαλιστικό τρόπο και ικανοποιεί έτσι και τους αντικειμενικούς στόχους ε, της οργάνωσης. Ευχαριστώ. Μιλούμε για τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Όπως έχουμε συζητήσει προ λίγων εβδομάδων, η ομάδα, η ΣΥΑΡΑ έχει την ίδια θέση και για τούτον εδώ τον κανονισμό, για την ΕΜΣΑ δηλαδή. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να τονίσω ότι προφανώς η συνεργασία αυτή με τροπολογίες στον κανονισμό δεν σημαίνει ότι θα λύσουμε έτσι όλα τα προβλήματα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ωστόσο ότι με τους δεδομένους πόρους, με την νέα αυτή συνεργασία, επιθυμούμε να σπρώξουμε τις χώρες εκείνες που είναι ιδίως εκτός Σέγγεν να συνεργαστούν. Διότι αν δεν κατορθώνουν να προστατεύσουν τα σύνορά τους από μόνες τους ε, και επειδή θέλουμε να διασώσουμε τον χώρο Σέγγεν, πρέπει να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί σημαντικά η ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε σωστή πορεία με την έκθεση που προτείνει η Επιτροπή. Εμείς εμένουμε βέβαια στην αρχή της επικουρικότητας. Είναι αρκετά ισορροπημένη από αυτή την άποψη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι αν μια χώρα μέλος ζητήσει ένα μηχανισμό μετεκαταστάσεως ή βγει εκτός Δουβλίνου θα πρέπει να δεχτεί τότε την υποστήριξη του οργανισμού και στη, να συμμετάσχει και η ΕΜΣΑ σε αυτή τη συνεργασία με τον οργανισμό. Δεν επιθυμούμε λοιπόν να καταθέσουμε τροπολογίες. Η ομάδα μας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών μπορεί να στηρίξει τις περισσότερες από τις τροπολογίες της εισηγήτριας. Αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε ότι η πρόταση της ε, Κομισιόν είναι ισορροπημένη και συμβαδίζει και με τους άλλους κανονισμούς για την εξωτερική φυλάξη των συνόρων. Εσάς Μπιλβάο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από την εισηγητρία. Γιατί είχα άλλη συνεδρίαση που δεν τελείωσε καιρός και δεν την άκουσα. Έχω όμω ε, το κείμενό της, το μελέτησα και έχω να πω το εξή. οργανισμός ΕΜΣΑ έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και είχαμε και πάρα πολλές συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι ένας οργανισμός στην οποία προσθέτουμε και πόρους και αρμοδιότητες πάντα σε οριακές καταστάσεις και ε, τελευταία στιγμή και όταν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, ε, όπως σε προκειμένο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια αφετηρία γιατί η ΕΜΣΑ είναι ακόμα ένας οργανισμός, ε, ένα μέσο που θα πρέπει να συνεργαστεί για να λύσουμε το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη. Αντίστοιχα όμως θα πρέπει να πω ότι εμείς δεν καταθέσαμε καμία τροπολογία ως ομάδα φιλελεύθερη, διότι δεν συμφωνούμε με την αιτιολογική έκθεση, ούτε τη γραπτή, ούτε το όσα ακούσαμε μόλις από την εισηγήτρια για όλα τα, αυτά τα ζητήματα του μεταναστευτικού εμείς πιστεύουμε ότι βεβαίως και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα της ασφάλειας, να βελτιώσουμε τον έλεγχο, αλλά σε αντίθεση με την εισηγήτρια, αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε αποκλειστικά ως απειλή, ούτε πιστεύουμε ότι είναι κάτι που έχει να κάνει με συναισθηματισμό. Είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα αυτό το οποίο οικοδομούμε και για μας το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει αρχές, ουσία, αξίες, που είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε ακόμα περισσότερο, αν γίνεται, σε περιόδους κρίσης παρά σε περιόδους που πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν συμφωνούμε ούτε με το κείμενο, ούτε με το ύφος, ούτε με την έκφραση, ούτε με την αιτιολογική έκθεση. Επιπλέον, για μας είναι απαράδεκτο να μας ε, ε, ε, αποδίδουν τέτοιες εκφράσεις ότι οι ηγέτες ε, των ε, κρατών μας ε, διοργανώνουν την αφέμαξη με επιδρομή των χωρών αυτών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες για να τους αφαιρούμε όλο το εργατικό δυναμικό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ούτε με τη συζήτηση έχει σχέση, ούτε με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό. Εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες και στο Σέγγεν, όπως σας είπα, και δεν συμφωνούμε για δύο βασικά πέρα από τα όσα ανέφερα προηγουμένως. Αυτή την εθνική εστίαση που θέλει να δώσει η φιλοδοξία συγκήτρια, γιατί από την οικονομική κρίση που ζήσαμε πριν από 4-5 χρόνια είδαμε ότι το να υπάρχουν ευρωπαϊκά εργαλεία, ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ε, και η δημιουργία τους μας έδωσαν λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά προβλήματα που γνωρίσαμε. Και προκειμένου, επίση δεν θεωρούμε ότι πρέπει να ορθώσουμε νέα σύνορα, γιατί δεν είναι λύση αυτό. Για άλλη μια φορά, βλέπουμε καθυστερημένη λύση και θέλω ότι Θέλω να ξαναθυμίσω ότι ε, με την κυρία Μάλστρομ είδαμε στην περασμένη θητεία όταν υπήρξε αυτή η τραγωδία της Λαμπετούσα πήγε την πρόταση στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο έλεγε ε, ή ε, μάλλον ε, υπενήχθηκε ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης αφορά μόνο την Νότια Ευρώπη. Και τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την ολιγορία γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όταν εμφανίζονται και τα προβλήματα, όχι όταν μας κατακλείζουν. Ο ΕΜΣΑ είναι ακόμα ένα εργαλείο για να δώσουμε μια λύση που θέλουμε και ανθρωπιστική αλλά και αλληλέγγυα είναι υποχρέωσή μας, τουλάχιστον εκείνων που θεωρούμε τον εαυτό μας δημοκράτη, που πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και πιστεύουμε στο μέλλον της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με αυτά τα είπε στην αρχή της παρέμβασής της εισηγήτριας για τους πρόσφυγες και την άποψη που έχει για την ανθρωπιστική κρίση. Εμείς αυτές τις εβδομάδες όλο στοιχείο συζητάμε την ένταξη στην αγορά εργασίας των προσφύγων και σε τεχνικό επίπεδο μας εξηγούν τι δυνατότητες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δεν χρησιμοποιούμε, θα και δεν είναι ενημερωμένα τα κράτη-μέλη για να τα χρησιμοποιήσουν και ότι υπάρχουν δίκτυα πόλεων που είναι διατεθειμένες να υποδεχθούν τους πρόσφυγες, αλλά αυτό δεν συμβαίνει γιατί τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τις, προς, τις ε, ποσοστούσεις τις οποίες καταρχήν είχαν ε, υποχρεωθεί να δεχθούν. Το να λέμε ότι θα πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί από την Ευρώπη προς όφυλος των Ευρωπαίων πολιτών είναι εντελώς απαραδέκτο διότι έχουμε υποχρέωση να παρέχουμε το δικαίωμα στο άσυλο Και δυστυχώς αυτό έρχεται μαζί με την πολύ αυστηρή πολιτική λιτότητα στην οποία υφίστανται οι ευρωπαϊκοί λαοί τον τελευταίο καιρό. Τώρα, ε, για την ακτοφυλακή, την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Η διαδικασία που επελέγει είναι ιδιαίτερος ταχεία, έκτακτη. Ε, δεν θα ήθελα να επιμείνω πάνω σε αυτό, αλλά είναι σαφές ότι αν πράγματι θέλουμε να καταλήξουμε σε συνεκτικές λύσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα πράγματα θα πρέπει να τα κάνουμε με διαφορετική μέθοδο και όχι με αυτή που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Τώρα, σε σχέση με την πρόταση έχουμε αρκετές διαφωνίες, αλλά ε, σε σχέση ε, η θέση η δική μας για την υπόθεση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην διαφάνεια, στον ξεκάθαρο χαρακτήρα του υλικού περιεχομένου της συνεργασίας που προβλέπεται. Στο κείμενο η συνεργασία αυτή δυστυχώς παρέχεται με πολύ θολό τρόπο, σε θεωρητικό επίπεδο είναι γεμάτη εφημισμούς η πρόταση, ενώ εμείς έχουμε να κάνουμε με ένα νομοθετικό κείμενο και περιμένουμε περισσότερα στοιχεία και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις ποια είναι τα ανώτατα όρια και ποιες είναι οι διαθεσιμότητες. Είναι λοιπόν απαραίτητο ότι ε, αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανεπαρκή. Τα θέματα της ασφάλειας στη θάλασσα στην ουσία αντιμετωπίζονται μόνο σαν θέματα ασφάλειας των συνόρων και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε δεύτερον τώρα σε σχέση με την εγγύηση των δημοκρατικών ε, ε, ιδεών. Ο εκτελεστικός ε, διευθυντής αυτή της ε, υπηρεσίας δεν εκλέγεται δημοκρατικά και έχει την απόλυτη εξουσία για να λαμβάνει αποφάσεις για την πολιτική διαχείριση του Frontex όπως ε, την άμεση επαναπροώθηση, τη χρήση βίας, ε, την υιοθέτηση συμφωνιών συνεργασίας με τρίτες χώρες και άλλα δεσμευτικά μέτρα. Τέτοιου είδους αποφάσεις, αν ληφθούν, θα πρέπει να είναι αποφάσεις οι οποίες θα έχουν με συνένεση ληφθούν, ληφθεί συγγνώμη, σε επίπεδο ευρωπαϊκό και δημοκρατικό. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει και η ξεκάθαρη έλλειψη σεβασμού και απόρριψη των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της διεθνούς ένομης τάξης ενώ είναι κάτι το οποίο ε, θα έπρεπε ε, να χαρακτηρίζει τον έλεγχο των συνόρων και την δημιουργία μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη να χορηγεί το άσυλο, να σέβεται το δικαίωμα του ασύλου και θα πρέπει να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να το κάνουμε. Και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε μια σωστή στρατηγική καταπολέμησης της σώματεμπορίας ή του τράφικινγκ αν θέλετε, Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πλειοψηφία των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιείται από τους μετανάστες είναι μαφιόζικου τύπου. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που πέφτουν στα χέρια ε, της μαφίας γύρω από τα σύνορά μας, που εκμεταλλεύονται την απελπισία των ανθρώπων αυτών, που στερούνται φυσικά και τις ελάχιστες ενημέρωσης. Συνεπώς λοιπόν εμείς θέλουμε να απορρίψουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως επίσης να απορρίψουμε και την έκθεση την οποία προτείνει η συγγήτρια. Για τους λόγους λοιπόν που έθεσα ε, νομίζω ότι το ελάχιστο που μπορούμε να απαιτήσουμε από μια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να σταματήσει να μην σέβεται ή να σέβεται όλο και λιγότερο τις δημοκρατικές αξίες ε, και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους του κοινωνικού. Ευχαριστώ πολύ. Keith Taylor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλά λοιπόν, συνάδελφοι, η συνθήκη των Ενωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, μιλώ για την συνθήκη του 1953, επιβάλλει υποχρώσεις στις χώρες να προσφέρουν δηλαδή καταφύγιο σε ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις χώρες τους εφόσον φοβούνται δίωξη για πολιτικούς, θρησκευτικούς ή και πολλούς άλλους λόγους. Μπορεί η και πολλους αλλους λογους μπορει η συγκιτρια να θεωρεί ότι ίσως τα Ενωμένα Έθνη δεν είναι κατάλληλα για να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Όμως να πω στις συναδέλφους μου ότι δόξα το Θεώ η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται παρόντες εδώ καταβάλουν προσπάθειες για να συμβάνουν στην επίλυση των προβλημάτων του κόσμου. Η συγγετριά χρησιμοποιεί το σχέδιο εκθέσεώς της για να προβεί σε πολιτικές δηλώσεις για ε, την έκθεση εννοώ δηλαδή για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ε, Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν, επειδή είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών, εν μέρη, και υπάρχει και άλλη δήλωση σε προηγούμενη γνωμοδότηση, αλλά δεν αναφέρεται εδώ σε ναυτιλιακή πολιτική. Αλλά αναφέρεται σε, όπως λέει, ακατάλληλες ή ανεπαρκείς ε, αντιδράσεις ή απαντήσεις στα προβλήματα της διακίνησης ε, προσφυγών και μεταναστών στην Μεσόγειο. Απολύτως απαράδεκτο και τυπικά και ουσιαστικά. Και γι' αυτό θα επιμείνω εμφατικά αυτή η εισηγητική της έκθεση να διαγραφεί. Προτείνει και οχτώ τροπολογίες η εισηγήτρια. Έξι από αυτές δεν αναφέρονται σε θέματα πολιτικής μεταφορών, αλλά σε διακρίσεις σε βάρος μεταναστών. Εμείς προτιθέμεθα να καταθέσουμε τροπολογίες επί της προτάσεως της Κομισιόν με στόχο να την βελτιώσουμε και θα καταψηφίσουμε το σύνολο της εκθέσεως που προτείνει η συγκήτρια. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νταμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά πρέπει να σχολιάσω, καλούμε να σχολιάσω την πρόταση της συναδέλφου του Εθνικού Μετόπου και αναγκάζομαι για μια ακόμη φορά να διαβάζω φράσεις οι οποίες είναι σοβαρά ελλειπτικές. Να τις ότι αυτό το οποίο θα σαν Επιτροπή δεν είναι να βρούμε την ευρωπαϊκή αντίληψη για την τρομοκρατία είναι κάτι το οποίο αυτή κάνει με πολύ υπεραπλουστευμένο τρόπο. Η πρόταση της Επιτροπής είναι ευρύτερη και σαν Επιτροπή Μεταφορών δεν πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε θέματα τα οποία διαφεύγουν των αρμοδιοτήτων μας. Ε, για μια ακόμη φορά λοιπόν στην ουσία εδώ ε, θα έλεγα οσμιζόμεθα στοιχεία κακώς εννοούμενου λαϊκισμού στα δηλώσεις της εισηγήτρια και το διαβάζω για να μην κάνω λάθος είναι ότι οι προσπάθειες που οργάνωσε η Ιταλία και που συντόνισε η Frontex ενθαρρύνουν ένα μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών να ξεκινούν για να έρθουν μέσα από επικίνδυνα δίκτυα στην Ευρώπη και έτσι ενισχύουν τους θανάτους, τα ναυάγια και, την, ε, και το τράφικινγκ. Μα πώς το λέτε αυτό, πώς επιτρέπετε στον εαυτό σας να το πείτε αυτό. Λέγατε ότι η Ιταλία προσελκύει την παράνομη μετανάστευση και τη σωματεμπορία. Αυτό είναι απαράδεκτο, άκερο, ανεπίκαιρο στο εσωτερικό μιας έκθεσης που θα πρέπει να εκπροσωπεί το σύνολο του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για τα στοιχεία που μας δίδετε και τα οποία γνωρίζουμε από το Frontex, από τον ΟΗΕ και τα λοιπά μιλώντας για πρόσφυγες. Βέβαια οι αριθμοί αυτοί είναι άνθρες και γυναίκες. Ένας πρόσφυγας είναι πρόσφυγας ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου και θα πρέπει να μας εξηγήσετε πώς μπορείτε να καθορίσετε εσείς ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος δεν είναι και φυσικά για να το κάνετε να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα. Και τέλος, ο παραλληλισμός που κάνετε ανάμεσα στη μετανάστευση και την τρομοκρατία είναι λαϊκιστικός, επικίνδυνος και ανακριβής. Το πρόβλημα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερος περίπλοκο και μετά από αυτά που έγιναν τον προηγούμενο μήνα θα έλεγα είναι κάτι που άπτεται βαθυτά των δυναμικών διαδικασιών που έχουν σχέση κυρίως τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες. Λοιπόν, ας μην λέμε τέτοια λόγια, ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τότε θα έχει νόημα να προτείνουμε τροπολογίες. Ας επανέλθουμε στο, ε, στην ουσία του θέματος. Στην ουσία της εκθέσεως. Δεν είναι και τόσο απλό. Και εκεί χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές και προσεκτικοί. Σε ό,τι αφορά την διεύρυνση δηλαδή του πεδίου εφαρμογή για, την, ε, για τις δράσεις της ΕΜΣΑ, ε, τίθεται κάποια ιδιαίτερα θέματα. Ανταλλαγή πληροφοριών. Και επίσης ανταλλαγή ή κοινή χρήση ε, υλικών και προσωπικού. Πολύ μακριά από την αρχική από, το αρχικό, από τα αρχικά καθήκοντα της ΕΜΣΑ. Λοιπόν, ολόκληρη η έκθεση δεν είναι και τόσο απλή, διότι ζητεί από τις χώρες μέλη να επανεξετάσουν τις νομικές τους θέσεις, είτε για τις ακτοφυλακές τους, είτε και για άλλα θέματα. Στην πρώτη έκθεση της κυρίας Ανωτή, την προηγούμενη φορά δηλαδή που συνέταξε έκθεση, είχα πει τότε ότι η θέση του Ενωμένου Βασιλείου, επειδή δεν συμμετέχουμε στο Σέγγεν, θα συνεργαζόμασταν, αλλά θα απήχαμε από την ψήφιση της έκθεσης. Εδώ είμαστε σε παρόμοια κατάσταση και λόγω των δύο αυτών χώρων. Όχι όμως μόνο το Ενωμένο Βασίλειο. Κάποιος έχει σταθεί μπροστά μου Ευχαριστώ που ε, απομακρύνετε. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τομείς κλειδιά που δεν αφορούν μονάχα το Ενωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλες χώρες μέλη. Άρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές και προσεκτικοί. Αντιλαμβάνομαι ότι στο Συμβούλιο συνεδριάζουν πολλές ομάδες εργασίας και συνεχίζεται μια εργασία για μια προσπάθεια επίλυση των θεμάτων αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να δω πώς εξελίσσεται η προσπάθεια αυτή πριν να συζητήσω περισσότερο. Και σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση ή μάλλον τις απόψεις της κυρίας Ανωτή, δεν συμφωνώ απολύτως ε, μαζί τη. Έχει όμω το δικαίωμα να εγείρει την φωνή τη στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή. Είδε μη, τη δημοκράτη είμαστε. μπορεί να μην ε, αντιδράσω απόλυτα στις ε, ε, παρατηρήσεις της αυτές, αν και μπορεί να έχω διαφορετικές απόψεις. Και πάντως χρειάζεται μια επικοδομητική συζήτηση. Υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε. Δεν θα υποστηρίξουμε απαραίτητα ορισμένες από τις τροπολογίες της, άλλες όμως δεν μας φαίνονται τόσο άσχημες και χρειάζονται και κάποιες ε, προσαρμογές. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να απευθυνθώ στην εισηγήτρια και να τη θυμίσω ότι η αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή, μάλλον ότι εδώ δεν είμαστε Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, είμαστε Επιτροπή ΤΡΑΝ, μεταφορών, όχι εσωτερικών. Άκουσα την εισαγωγή της και φοβάμαι ότι δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται, να τα ξαναπώ μήπως. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, ε, εγώ έχω κριτική στάση απέναντι στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε μια στάνταρτ ε, αντίδραση στην Ευρώπη. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι. Ε, και για να γίνει κάτι εκχωρείται και άλλη εθνική κυριαρχία και εγώ δεν είμαι σύμφωνος με αυτά. Ακούμε να γίνεται λόγος και για ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Αυτό είναι πάρα πολύ παραπλανητική πρόταση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ούτε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, ούτε λιμενικό σώμα, ούτε πρόκειται να έρθει. Είναι οργανισμοί μεταξύ αυτών Frontex και Emsa, και εθνικές ακτοφυλακές που συνεργάζονται. Έτσι δεν είναι. Ε, μπορούν να υποστηριχθούν, να δεχθούν βοήθεια στις δράσεις και δραστηριότητες ε, στην διάσωση προσφύγων. Αλλά Άλλο πράγμα είναι να θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Υπό την έννοια αυτή, Πρόεδρε, συμφωνώ με τις επικρίσεις της ηγήτριας ε, και θα κάνω και σχετικά τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Ιζαμπέλα Δεμόντε. Sì, grazie. Ε, anche da parte mia devo dire c'è και εγώ δεν μπορώ παρά να διαφωνήσω με την πρόταση της κυρίας Αρνοτού λόγω κυρίως των αιτιολογικών σκέψεων. Είναι στην ουσία μία πρόταση η οποία ζητά τη μη έγκρισή της διότι αμφισβητεί τους πυλώνες της ίδιας της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο στρέφεται κατά της βάσης της ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών και όπως εξήγησαν και άλλοι συνάδελφοι δεν υπάρχει, δεν είναι η πρόταση που γίνεται μια πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών. Περιλαμβάνει επίσης επιπλέον στοιχεία τα οποία είναι απαράδεκτα, αναφέρεται στους πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται εδώ με τεράστιους κινδύνους για τη ζωή τους και δίδει στην προσπάθειά τους αυτή ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο και όπως είπε και η συνάδελφος Νταμάτο σχετικά με αυτά τα οποία έχει κάνει η Ιταλία με το Mare Nostrum η Ιταλία και το Frontex ε, δεν έχουν ενθαρρύνει την άφηξη των μεταναστών είναι μια πρόκληση αυτή την οποία θεωρώ ε, μη γενναιόδορη και προκλητική απέναντι σε αυτούς οι οποίοι απλά προσπαθούν να σώσουν ζωές ανδρών, γυναικών και παιδιών. Και δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε να χαθούν αυτούς τους ανθρώπους. Και η ταύτιση τώρα μετανάστευσης και τρομοκρατίας είναι μία από τις ε, κλασικές λαϊκίστικες δηλώσεις που ακούμε στην Ευρώπη. Η πραγματικότητα διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς σχετικά ε, με την προέλευση των τρομοκρατών που είναι πολλές φορές τρίτη και τέταρτη γενιά Ευρωπαίων πολιτών. Σχετικά τώρα με το περιεχόμενο το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει η ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, η αποκατάσταση των συνόρων μόνο ευνοϊκή δεν είναι για την επίλυση του προβλήματος, ε, και είναι κάτι που λειτουργεί και εις βάρος ε, των εμπορικών συναλλαγών. Ας πούμε στον τομέα ε, των οδικών μεταφορών καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι μία ώρα αναμονής θα έχει 40 εκατομμύρια ζημία προκαλέσει. Ευχαριστώ, Ντομινίκη, και Δύο λόγια μόνο, Πρόεδρε ως Γάλλος ε, σημείωσα ιδιαίτερα αυτά που είπε η κυρία Γνούτση. Δεν θέλω να επανέλθω στα όσα υπόθηκαν. Συμφωνώ με πολλά για τους ε, μετανάστες, ε, τα χαρακτηριστικά τους που είναι εκτός ε, θέματος. Κάτι άλλο που μας προκαλεί έκπληξη. Το γενικό ύφος της έκθεσης κυρίας Αγνοτσού είναι να μας εξηγήσει ότι αυτό που χρειάζεται τελικά είναι να ενισχυθεί η επικουρικότητα, δηλαδή η εθνική κυριαρχία των κρατών μελών ε, για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στον έλεγχο της μετανάστευσης. Δεν θα μπω τώρα στη συζήτηση. Συμφωνώ με τα σχόλια ε, για το άσυλο και τους πρόσφυγες. Ως εδώ όμως ε, διαφυλάσσεται απολύτως ε, κυρία Αγνωτή η εθνική κυριαρχία. Δεν υπάρχει καθόλου ευρωπαϊκή συνεργασία γιατί δεν έχουμε χωρίσει κυριαρχία για τα σύνορα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή φυλακή διότι θα αντιτίθεται αυτό στις συνθήκες. Ε, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες και μέσα της Frontex που δόθηκαν στη διάθεση κάποιων χωρών τελείως γελία σε σχέση με τις ανάγκες. Γι' αυτό που λέτε μάλλον που δεν λέτε είναι ότι θα πρέπει να, ενισχυθεί ο έλεγχος στο σύνορο με περισσότερη κυριαρχία εθνική και καθμία ε, ευρωπαϊκή συνεργασία. Θέλω να υπενθυμίσω στην εισηγήτρια ότι οι χώρες που σήμερα υφίστανται μεταναστευτικέ ε, πιέσει είναι ορισμένε. μόνο. Δεν άκουσα εγώ η Δανία ή οι κάτω χώρε να υφίστανται τεράστιε μεταναστευτικέ πιέσει στα σύνορά του. Οι χώρες εκείνε λοιπόν που υφίστανται τεράστιε πιέσει, δεν δίνονται να ανταποκριθούν, δεν έχουν τα μέσα μόνες του. η ενίσχυση της κυριαρχίας θα τις άφηνε αντιμέτωπες ε, ενώπιον των ευθυνών τους και η κατάσταση που γνωρίζω θα ήταν ακόμα πιο ε, σοβαρή. Είναι λογικό λοιπόν και επόμενο η Ευρώπη να τρέξει να βοηθήσει τις χώρες που έχουν αυτό το πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και μόνο με συνένωση των ευρωπαϊκών ε, μέσων και με χώρες κυριαρχίας μπορούμε να βρούμε λύση ε, σε αυτό το πρόβλημα. Στην Ελλάδα ε, οι ε, εθνικές αρχές έχουν ε, απολύτω ξεπεραστεί από τι εξέλιξει. Δεν έχουν χώρισει καμία εθνική κυριαρχία. Βεβαίω πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Αλλά αν αφαιθεί στα χέρια των κρατών μελών, πράγμα που ισχύει σήμερα, έχει τεράστιε ελλείψει. Η κοινοτική μέθοδος νομίζω είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, Μπάρμπαρα Σεδιέ, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Αρμόδιας ε, Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εάν με επιτρέπετε, θα επικεντρώσω τις παρατηρήσεις μου στις ναυτιλιακές μεταφορές και στην πρόταση για την ΕΜΣΑ αν και η συζήτηση σας επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα σήμερα. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για την ΕΜΣΑ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν πρόκειται μόνο για έλεγχο των συνόρων. Πρόκειται συνολικότερα για την ενίσχυση της συνεργασίας για τα καθήκοντα ακτοφυλακής. Αυτή η ανάγκη ενισχυμένου συντονισμού αναγνωρίζεται και στη νέα νομοθεσία στην οποία συμμετέχει ως νομοθέτης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρεται αυτό και στο προήμιο αλλά και στη έκθεση για τις προσπάθειες καταπολέμησης της ρήπανσης. Και η έκθεση της Επιτροπής το 2014 που σημείωνε τα αποτελέσματα της έλλειψης συνεργασίας ακτοφυλακών στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΕΜΣΑ, αυτή υποστηρίζει ήδη τις ε, δραστηριότητες ακτοφυλακής των χωρών μελών για μέτρα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η πρότασή μας έχει τον στόχο να εξασφαλίσει ότι η ΕΜΣΑ θα συνεργαστεί με την ΕΦΚΑ και με την Frontex για να χορηγήσει υποστήριξη στις χώρες μέλη, χωρίς να αλλάξει το πεδίο αρμοδιοτήτων των ε, οργανισμών αυτών. Τώρα, το κείμενο του άρθρου είναι το ίδιο και στην πρόταση Frontex και στην πρόταση ΕΦΚΑ. Μιλούμε για την ανάγκη διασφάλισης συνεργασίας των οργανισμών, την προώθηση συνεργειών στην υποστήριξη και στις υπηρεσίες που προσφέρουν στις χώρες μέλη σε διάφορους τομείς. Η ΕΜΣΑ κάνει ήδη πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την ναυτική εποπτεία, με την, ε, την ναυτική επιτήρηση, ε, με ένα προπολογισμό ο οποίος αφιερώνεται σε αυτό. Τέθηκε και μια ερώτηση για τους πόρου προηγουμένω. Ο προπολογισμό είναι της τάξη των 85 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια. Πολλά χρήματα δηλαδή σε σύγκριση με τον υφιστάμενο προπολογισμό ε, ΕΜΣΑ. Επίσης και προσωπικό. Επιθυμώ να ε, αναφέρω ακόμη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το 2016 για την συνεργασία δηλαδή των οργανισμών σε άσκηση καθηκόντων ακτοφυλακής. Και τέλος, επιτρέψτε μου να εξηγήσω ότι στην ουσία πρόκειται για μια προσπάθεια να βελτιστοποιήσουμε την χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, χωρίς να αλλάζουμε τίποτα σε ό,τι αφορά την διοίκηση των οργανισμών αυτών και σε ό,τι αφορά την έμσα, καμία αλλαγή σε αρμοδιότητες, ούτε ένταξη στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, καθηκόντων ακτοφυλακής. Μάλιστα, η κυρία Αρνοτού ε, και πάλι ως εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για τον πρώτο μιλητή, ο κ. κάμπ μας είπατε ότι οι αρμοδιότητες είναι των εθνικών κρατών, αλλά λέτε κάτι το αναλυθές, κάνοντας ότι δεν κάνω τη διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που ζητούν άσυλο και τους υπολείπους. Λάθος σας. Πρέπει να ξαναδιαβάσετε την παρέμβαση την οποία έκανα γιατί θα διαπιστώσετε ότι κάνω την διάκριση αυτή. Πολλοί κάνουν άλλωστε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτούς ε, ετούνται πραγματικά άσυλο και σε αυτούς που δεν είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Δεν... Ε, Grande différence entre la politique d'immigration qu'effectivement je combats ε, η πολιτική της μετανάστευσης είναι κάτι το οποίο καταπολεμώ, έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά ταυτόχρονα νιώθω, θα έλεγα, άσχημα για αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους κάνουμε να πιστεύουμε ότι το, η Ευρώπη είναι ένα ελντοράδο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν κατανοήσατε αυτά τα οποία σας είπα. Λέτε εσείς ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτά τα εσωτερικά σύνορα, εδώ διαφοροποιούμεθα γιατί εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Και άλλωστε και πολλοί συνάδελφοί σας από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Γαλλία συμφωνούν απολύτως με την δική μου άποψη. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο κύριος, ο Μιζελιέ, γιατί είναι αντιπρόεδρος μιας πολύ μεγάλης περιφέρειας και έχει εκφράσει τις αμφιβολίες του για το χώρο Σέγγεν. Συνεπώς λοιπόν πιστεύω και το λέω αυτό όλος μεγαλύνει. Δεν ακούμε την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών. Αν συνεχίσουμε να μην τους ακούμε, τότε πραγματικά τα προβλήματα θα είναι αξεπέραστα. Εσείς δεν θέλετε να αναφερθείτε στις Ισλαμικές τρομοκρατικές ενέργειες στη Γαλλία και στο Βέλγιο, αλλά απέδειξαν ότι το Σέγγεν δεν είναι βιώσιμο. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια σαφής αντίληψη που εδραιώνεται εναντίον αυτής της πολιτικής στην Ευρώπη. Και θυμίζω εδώ την, το εξαιρετικό εκλογικό αποτέλεσμα των φίλων του FPU στην Αυστρία. Θα ήθελα να απαντήσω επίσης και στην κυρία Άντερσον, τον κύριο Τσίλερ, και την κυρία Μπαραντίκα γιατί με κατηγόρησαν για τα ίδια πράγματα. Το ίδιο και η κυρία Γκονσάλες, ο κύριος Τέιλορ και η κυρία Νταμάτο. Με κάποιες βέβαια διαφοροποίησεις και να σταθώ σε αυτά που είπε η κυρία Νταμάτα, γιατί πραγματικά να αναλέτε ότι αυτό το οποίο μεταφράστηκε τουλάχιστον από τους μεταφραστές, ότι αποπνέω θα έλεγα την δυσοδεία του χειρότερου λαϊκισμού, είναι απαράδεκτο και δεν το δέχομαι και δεν είναι τρόπος αυτός άσκησης της πολιτικής. Λέτε ότι ένας πρόσφυγας είναι πρόσφυγας, αλλά πέραν τούτου ε, δεν βοηθάει και δεν θα απαντήσω στις ύβρις σας και δεν με ενδιαφέρουν οι ύβρις σας. Πολλοί από εσά αναφέρονται στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε ότι στιγματίζω τους μετανάστες, ότι δεν σέβομαι τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας και τη σεβόμεθα. Εγώ δεν το πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Μου λένε επίσης ότι ε, δεν θα καταθέσει η κυρία Μπαραντίκα ε, τροπολογίες γιατί δεν συμμερίζεται την αιτιολογική έκθεση. Κοιτάξτε κύριε Μπαραντίκα, προφανώς διαφωνείτε με την αιτιολογική έκθεσή μου, με αυτά που σας είπα. Αλλά λέμε ότι η βασική αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ένωσης είναι ακριβώς ο σεβασμός της δημοκρατίας και του δημοκρατικού ελέγχου και δεν σας βλέπω να είστε πολύ δημοκράτης σε σχέση με αυτή την έκθεση και να θέλετε να γίνει συζήτηση εκτός από την κυρία Φώστερ η οποία πάντα έμφυση λογικής στις συζητήσεις. Λοιπόν, μου λέτε ότι δεν είναι παράλογο να μην υποδεχθούμε τους μετανάστες. Κύριε Τέιλορ, είπατε ότι δεν ψάχνουμε εμείς να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Δυστυχώς αυτό είναι το λάθος που κάνουμε και εσείς κυρίως κάνετε. Σας προανέφερα αυτά που είπε ο Ντόναλτ Τάσκο, ότι ένα από τα προβλήματα της Ένωσης είναι ότι προσπάθησε να λύσει τα προβλήματα του κόσμου χωρίς να λύσει τα προβλήματα της Ένωσης. Λυπάμαι λοιπόν γιατί δεν μπορούμε όπως είπα να κάνουμε μια συζήτηση ειρηνική. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα αυτό θα προκαλέσει επιπλοκές. Εσείς πιστεύετε ότι απαιτείται περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, λιγότερα ευρωπαϊκά σύνορα. Ζείτε στην ουτοπία ότι τα εξωτερικά σύνορα θα προστατεύσουν τους πολίτες μας. Όχι, αυτό δεν θα γίνει, δεν το πιστεύω. Και νομίζω ότι για μια τέτοια έκθεση θα έπρεπε να είναι κανείς λίγο πιο ψύχρεμος και να σεβαστεί λίγο περισσότερο τις απόψεις ημέν δε. Γιατί εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι παρόλα αυτά όλοι εδώ έχετε έρθει για να εκφράσετε τις απόψεις των πολιτών σας δεν εξελέγει με μέσω της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς λοιπόν σε ό,τι αφορά στη Γαλλία, εγώ ήρθα εδώ για να προστατεύσω την ασφάλεια των πολιτών μου. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμός ε, της γνώμης του άλλου δεν είναι μονόδρομος, ξέρετε, είναι διπλής κατεύθυνσης. Λοιπόν, προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 28 Απριλίου στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης Ευρωπαϊκή Στρατηγική για ε, το χώρο των Άλπαιων με εισηγήτρια την κυρία Αγιώτο η οποία απουσιάζει και θα την εκπροσωπήσει η κυρία Νταμάτο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ αντικαθιστώ εδώ την κυρία Αγιούτο η οποία έχει παραμείνει στην χώρα της ε, λόγω ενός απρόβλεπτου συμβάντος. Θα ήθελα λοιπόν εξ ονόματος της κυρίας Σαγιούτο να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εξαιρετική δουλειά την οποία έκαναν στη συνάντηση των σκιωδών την προηγούμενη εβδομάδα. Τους ευχαριστώ για τον επικοδομητικό διάλογο κατατέθηκαν 94 τροπολογίες. Εμείς προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε συμβιβαστικές προτάσεις. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρότειναν οι συνάδελφοι με βασικό στόχο το να διατηρηθεί μια περιοχή η οποία λόγω της γεωμορφολογικής της εικόνας είναι ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη στον τομέα του περιβάλλοντος αλλά και των ευρωπαϊκών μεταφορών. Πολλά είναι τα επιχειρήματα τα οποία συζητήθηκαν μέχρι τώρα. Θυμίζω το θέμα του τουρισμού και την δυνατότητα εκμετάλλευσης του δυναμικού της περιοχής, να ξεπεράσουμε την εποχικότητα και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να βελτιώσουμε την συνδεσιμότητα ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές με πολλές μορφές μεταφοράς και μέσω των κοινοτικών ταμείων και εκμεταλλευόμενοι υπάρχοντα δίκτυα. Να ενθαρρύνουμε το λεγόμενο shift to rail Νομίζω ότι επίσης πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις υδρολογικές ενεργειακές ικανότητες και να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Σημαντικό είναι να δούμε τι γίνεται με τις, διαμεθο... με μεθοριακές περιοχές. Εδώ θα έλεγα να μην αγνοήσουμε την κατάσταση των μεταφορών στην περιοχή, να δούμε ε, πού χρειάζονται επενδύσεις, και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε και τη συνδεσιμότητα την τοπική προστατεύοντας το περιβάλλον. Η επόμενη συνάντηση των σκιωδών θα γίνει την 12η Μαΐου στο Στρασβούργο. Ας φέρουμε κοντά λοιπόν τις θέσεις μας για να στηρίξουμε ένα τελικό κείμενο το οποίο θα το δεχόμαστε όλοι. Εμείς θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να προσφέρει στην διαμόρφωση της τελικής έκθεσης με σωστό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κλάουντια Σμιτ. Ευχαριστώ. Τώρα είναι δύσκολο όταν ε, ε, κανείς απουσιάσει από τη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών, αυτά που είπατε εγώ δεν τα άκουσα σε εκείνη τη συνεδρίαση, εν ε, τι έχει σημασία σε αυτή την έκθεση οι αποφάσεις στην πολιτική μεταφορών να συνδιαμορφώνουν ε, τις αποφάσεις και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που έχουν και άλλοι τομείς πολιτικής. Εδώ πρόκειται για υποδομές ε, που έχουν επιπτώσεις ε, χρόνια ολόκληρα και δεκαετίες. Καλό θα είναι λοιπόν κάπως σοβαρά και ευσυνείδητα να δουλεύουμε. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα επιβαρύνει το χώρο των Άλπαιων από τις μεταφορές γιατί υπάρχει άξονας βορράς νότος ε, από τα διάσελα και τις διαβάσεις των Άλπαιων και είναι, ε, αυτό και αφετέρου είναι βαριές υποδομές και δαπανηρές. Μία από τις βασικές προκλήσεις λοιπόν είναι ο χώρος των Άλπαιων να διαφυλαχθεί ως ένας χώρος όπου ζει κόσμος και ε, προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος θα πρέπει αφενός να είναι μέλημά μας αφετέρου ε, και ε, να ανθίσει και να αξιοποιηθεί, να υπάρχει δυνατότητα για σύγχρονη ζωή και οικονομία. Γι' αυτό χρειάζονται συνδέσεις της περιοχής των Άλπαιων με τις, τα πρωτεύουσες και τα άλλα μητροπολιτικά κέντρα. 46 περιφέρειες αυτοοργανώνονται και αυτοδιοικούνται για να λύσουν τα προβλήματα. Αυτό είναι χαρμόσυνο και το καλωσορίζουμε. Αλλά αυτή η διάσταση δυναμητίζει τις δυνατότητες ε, της περιφέρειας. Ξέρουμε ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα έχουν πρόβλημα χρηματοδότησης. Μέχρι το 2020, 30 και 50 ακούμε διάφορα νούμερα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ε, εκπροσωπούνται σε πραγματικό ε, προϋπολογισμό, αυτά που κυκλοφορούν. Θα χρειαστούν τεράστιες ε, προσπάθειες από τα κράτη-μέλη και από τις περιφέρειες για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Και αυτά τα δίκτυα έχουν και ένα συμβολικό χαρακτήρα για την οικοδόμηση της Ευρώπης και ε, την ολοκλήρωση, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Κάτι άλλο που είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι χρειαζόμαστε αξιόπιστες συνδέσεις μεταφορών και συγκοινωνιών για την οικονομία μας και όσο γίνεται περισσότερο φιλικές στο περιβάλλον. Εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή και τα μέσα στις περιφέρειες για να φτάσουν σε αυτό το στόχο, ενώ και τα οικονομικά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, να ε, ε, ε, χτίσουν αυτές τις υποδομές, αλλά και τα επιχειρήματα για να υπάρξει αποδοχή επιτόπου. Το λένε και κάποιες τροπολογίες. Ε, όλοι ε, οι δήμοι, κοινότητες, πολίτες, ΜΚΟ έχουν την ε, δυνατότητα, έχουν και το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαβούλευση. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε η μετάβαση στο σιδηρόδρομο. και κάποιοι θέλουν να καταρρύψουν ε, αυτό το επιχείρημα υπέρ του σιδηροδρόμου για λόγους υπερβολικής παρέμβασης στη φύση. Όποιοι απαιτούν μόνο, χωρίς να δίνουν ε, ε, τη δυνατότητα υλοποίησης όλων αυτών και την ηλική και την οικονομική, δεν λαμβάνουν τελικά σοβαρά υπόψη. Θα πρέπει να έχουμε τη μεγαλύτερη ελευθερία για τους πολίτες, ε, για τις επιχειρήσεις, ε, διαφυλάσσοντας όσο γίνεται περισσότερο το περιβάλλον και τη φύση. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Τώρα με ποια μέσα θα φτάσουμε σε αυτό το σκοπό. Αυτή είναι η δουλειά μας και να μην υπερφορτώνουμε τώρα αυτό το σχέδιο με άλλα άσχετα πράγματα που δεν έχουν και σχέση με τη δική μας Επιτροπή Μεταφορών. Ε, έγινε μια πρώτη συνεδρία των σχεδόν εισηγητών. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Αλλά εγώ επειδή είμαι εκφύσεως αισιόδοξη πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα αισιοπέρας από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Ιζαπέλα Ντεμόντα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Είχα μία συνάντηση σε επίπεδο σκιωδών και κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης η συγγήτρια είπε ότι θέλει να συλλέξει στοιχεία και να καταλήξει σε μία συνενετική πρόταση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ήδη από τη δεύτερη συνάντηση θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία για τα ακαθόδη προβλήματα πάνω στα οποία οι συζητήσεις ε, ήταν μέχρι τώρα έντονες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποιος είναι ο τελικός στόχος, ότι το κοινό πρόβλημα στις Άλπεις είναι η απίσχναση του πληθυσμού. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι συνέπειες έχει αυτό και ε, σε επίπεδο οικολογικό και ενδιαφέρομαι εγώ για αυτό το θέμα γιατί προέρχομαι από την αλπική περιοχή και να δούμε τι δυνατότητες αναπτυξιακές έχει η μεγάλη αυτή περιοχή. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν να δούμε και τι λέγει η σύμβαση για τις Άλπες, για τις Άλπες και τα πρωτόκολλα ανάπτυξης των μεταφορών και του τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις εδαφικές δικαιοδοσίες, γιατί το θέμα είναι να αναπτυχθεί η ορεινή περιοχή και όχι τόσο η, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τα μέσα για να το πετύχουμε αυτό, δηλαδή τις τοπικές διασυνδέσεις, θα πρέπει να υπάρξουν διασυνδέσεις και σε τεχνολογικό επίπεδο και με ευχαρίστηση άκουσα στην εισαγωγή ε, μια συγκεκριμένη αναφορά στον τουρισμό που είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και για την καταπολέμηση του εποχιακού χαρακτήρα της απασχόλησης που οδηγεί στην έλλειψη οικονομικής αηφορίας με, σχετικά τώρα με τα ten ε, Η αλπική περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή πυκνότητα υποδομών και μηχανοκίνητων μεταφορών και ε, διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και τέτοια δίκτυα είναι μεν αναπόφευκτα και δεν είναι θα έλεγα ασύμβατα με την δυνατότητα ύπαρξης ε, μιας τοπικής συνδεσιμότητας. Γιατί για να μπορέσει κανείς να, να... να, να ζήσει σε μια τέτοια περιοχή πρέπει να μπορεί να πηγαίνει με ε, ασφαλή τρόπο στον χώρο εργασίας του, και να μπορεί επίσης να εργάζεται και με τις νέες μορφές χωρίς να μετακινείται καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ζήλε. Δεν θέλετε. Σάσκουν Ευχαριστώ πολύ, Και εγώ θέλω να αρχίσω με ευχαριστίες προς την εισηγήτρια για το επικοδομητικό της πνεύμα. Συνεδρίασαμε την περασμένη εβδομάδα και ηγητές, 20 συμβαστικές προτάσεις μας ε, ε, κατέθεσε και κάναμε και βήματα πρόοδου σε πολλές. Οι δικές μας τροπολογίες έχουν εσωματωθεί σε συμβαστικές και κυρίως αφορούν την ενίσχυση ε, της ανάπτυξης της ψηφιοποίησης των ΚΙΚ για να υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα και η ψηφιακή και η διασύνδεση με τη νέα ψηφιακή εποχή. Και την περιφέρεια αυτή αυτό είναι εργαλείο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Άρα πολλές από τις τροπολογίες μας έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των ε, εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των κοινωνικών που δεν συμμελαμβάνουν για να μπορεί ο κόσμος να εκπαιδεύεται, να καταρτίζεται σε ποιοτικέ θέσεις εργασία και να εγκαθίστανται κιόλα αυτή την περιφέρεια που πλήττεται όπως και άλλες από, από ψήλωση. Υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες έτσι λοιπόν και στη συνεδρίαση είπαμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τα πριν από τρία χρόνια όταν κάναμε αναθεώρηση των ε, δικτύων και των, των προγραμμάτων ε, προτεραιότητας με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλειπε ακόμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αυτό το στοιχείο. Και θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το θέμα και να υπάρξει ε, κατάλληλη χρηματοδότηση από τη διευκόλυνση συνέοντας στην Ευρώπη. Είμαστε σε καλό δρόμο, ποντάρουμε εμείς σε αυτή τη στρατηγική για τις Άλπεις και να πριτανεύσει αυτό το επικοδομητικό πνεύμα της ηγήτριας για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και να βελτιώσουμε όλοι μαζί την αρχική πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Κίλιονεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια καθώς και όλες και όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν. Χρειαζόμαστε μια κοινή στρατηγική διότι η περιφέρεια ε, που θίγεται προκειμένου είναι μεγάλη και τα περιβαλλοντικά προβλήματα οφείλουν να λυθούν υπόψη. Το ίδιο όπως και ο τουρισμός για να προωθηθούν τα θέματα και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες. Επίσης, θεωρώ ότι επειδή οι κυκλοφοριακές ροές είναι μεγάλες και οι ανάγκες επίσης, οι επενδύσεις τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ υψηλές. Άρα, τα κεφάλαια που θα επενδυθούν πρέπει να επενδυθούν με τρόπο αποτελεσματικό, αποδοτικό. Με τρόπο ευφυή δηλαδή και σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των κατοίκων της ε, περιοχής. Ευχαριστώ, λέει ο ε, πρόεδρος η κυρία Αρνοτού. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, έχουμε καταθέσει μια τροπολογία Α, για, ναι, για τη γραμμή Λιών ε, Τουρίνο. Τωρίνο. Εμείς Έχουμε επίσης ε, προτείνει και μια τροπολογία για τις λευκές ζώνες. Μου φαίνεται κάπως παράξενο να μην λαμβάνονται υπόψη, Ιδίω βέβαια σε μια τέτοια έκθεση. Ευχαριστώ. κύριε Τέιλορ. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Ο συνάδελφό μου που δεν είναι παρόν σήμερα μου ζήτησε να πω ότι οι τροπολογίες που προτείνονται είναι καλές και τις δεχόμαστε. ενώ τον Ντάβορ Σκέρλετ. Και σωστό να τα υποστηρίξουμε όχι μόνο το ε, Μνημόνιο συμφωνία, αλλά και την ε, Σύμβαση των Άλπιων που έχουν κυρωθεί από την Ένωση και από τις ε, φυγόμενες χώρες μέλη να αναφερθούν και τα έργα για τις μεγάλες σύραγγες, θετικά μάλιστα. ο Μπρένερ και ε, η σύνδεση Λιών Τουρίνου. Ο βιώσιμος τουρισμός, για παράδειγμα ο συνδυασμός σιδηροδρόμου και ποδηλάτου, ε, είναι ένα στοιχείο που έχει μεγάλη σημασία και θα προσφέρει ε, και αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην περιοχή των Άλπων. Αυτά ήθελα να σας μεταφέρω. Ευχαριστώ. Ε, μου αρέσει πολύ αυτή η στρατηγική για τον χώρο των Άλπαιων και βλέπω να ανοίγονται μεγάλες δυνατότητες για το σύνολο της ε, περιοχής. Χρειάζονται κίνητρα, χρειάζονται οθήσεις για για το επιχειρηματικό δυναμικό αλλά και για την οικολογία. Μεγάλο δυναμικό ανοίγεται για αστικά και μη κέντρα. Εμένα με ενδιαφέρουν βέβαια ιδίω οι περιοχέ τη υπαίθρου και απομακρυσμένε περιοχέ, γιατί εκεί όλο και περισσότερο εγκαταλείπει ο κόσμο τι περιοχέ αυτέ και μεταβαίνει στα αστικά κέντρα. Επομένω ε, λείπει πια μια ισορροπία. Είναι σημαντικό λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αυτές προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό για την κινητικότητα, για τις διασυνδέσεις. Χρειάζεται λοιπόν να ε, ενισχυθούν τα δίκτυα μεταφορών και να υπάρξουν ασφαλείς και άνετες διασυνδέσεις, ώστε να ε, δοθεί και μια ποιότητα στην διαβίωση και των ανθρώπων. Φλόριαν Νάστ από τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο. Ευχαριστώ και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευχαριστώ την εισηγήτρια δηλαδή, αλλά βεβαίως και για τα σχόλια που έχετε κάνει και για την μακροπεριφερειακή προσέγγιση για τις Άλπεις. Μεταφορές και τουρισμός παίζουν κρίσιμο ρόλο για την περιοχή αυτή. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα πράγματα, τα οποία βέβαια ήδη λέχθηκαν σήμερα, από τη μια μεριά θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η στρατηγική αυτή απορρέει από την επιθυμία των περιφερειών και των χώρων μελών. Οι περιφέρειες βέβαια έπαιξαν εδώ ένα κέριο ρόλο προωθώντας την στρατηγική αυτή και αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Δηλαδή η στρατηγική αυτή δεν επιβάλλεται άνωθεν από το ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά είναι μια προσέγγιση από κάτω και αυτό φαίνεται καθαρά και από την αρχή της προσέγγισης αυτής. Ένα ε, πράγμα τώρα το οποίο καθιστά ιδιαίτερο το χαρακτήρα της θετικής αυτής είναι ότι για πρώτη φορά αυτή ασχολείται με ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο. Δηλαδή που περιλαμβάνει και όρείνες περιοχές αλλά και περιαλπικές. Μας ανοίγεται λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και αυτό βέβαια να μην το λησμονούμε όταν εγκύπτουμε στη στρατηγική αυτή, ότι δεν αφορά δηλαδή μόνο ορεινές περιοχές, ούτε μόνο μητροπολιτικές περιοχές, ούτε μόνο τις περιαλπικές περιοχές, αλλά ότι θα πρέπει να λειτουργήσει για τη νέα αμοιβαία ωφέλεια όλων αυτών των περιοχών, η οποία μάλιστα είναι και ευρύτερη από αυτήν που καλύπτει η, σύμβα... η συνθήκη των Αλπιών. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφερθεί και αυτή η Alpine Convention στην έκθεση, αυτό θεωρείται δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θα πρέπει να μην ότι πρόκειται για την καρδιά των Άλπαιων. Και ούτω ή άλλω το κείμενο τη συνθήκη είναι ήδη υποχρεωτικό. Ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης. Στη συζήτηση αυτό αναφέρθηκε σήμερα. Γνωρίζετε ότι δεν διατίθεται νέα κονδύλια για τις στρατηγικές αυτές, ούτε για τη μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις. Είναι πιο σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι υφιστάμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες σε τρόπο ώστε να εξυπηρετήσουν την ιδέα και τους στρατηγικούς στόχους της ε, προσέγγισης αυτής. Και βέβαια και από τα κονδύλια της, του Στρατηγικού Ταμείου Επενδύσεων, δηλαδή του Ταμείου Juncker. Αλλά βέβαια και η παραδοσιακή χρηματοδότηση από άλλες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ε, το Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως, τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, που είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων. Άρα, νομίζω ότι όλες και όλοι θα πρέπει να συμπαραταχθούμε στην προσπάθεια αυτή, έχοντας υπόψη βέβαια ότι και η επόμενη χρηματοδοτική περίοδος, το επόμενο δηλαδή πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα αρχίσει να γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και βέβαια οι στόχοι της αλπικής στρατηγικής θα απηχούνται στην ε, χρηματοδοτική αυτή στρατηγική. Ευχαριστώ λοιπόν ιδίως το Ευρωκοινοβούλιο ε, ιδιαίτερο μάλλον το Ευρωκοινοβούλιο και ιδίω στην Επιτροπή σας, η απόψει της οποίας θα βρουν απήχηση και στην τελική έκθεση της Επιτρόπου μου. Μάλιστα. Ρόζα Νταμάτο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εξ ονόματος της συναδέλφου Αγιούτο ε, οι προτάσεις της έγιναν ήδη, ελήφθησαν ήδη υπόψη και γι' αυτό στις 12 Μαΐου στην επόμενη συνάντηση η συζήτηση θα είναι ιδιαίτερος παραγωγική. Ευχαριστώ πολύ. Χρονοδιάγραμμα. Ψηφίσουμε στις 24 Μαΐου εδώ στην Επιτροπή μας. κομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω μόνο να κάνω μια μικρή διόρθωση γιατί στο τέλος ε, μίλησα για τη στρατηγική για το χώρο των Άνθεων αντί να πω των Άλπαιων, γιατί είναι η επόμενη συνεδρίαση που έχω και μου ξέφυγε. Εννοούσα ε, των Άλπαιων προφανώ και όχι τον Άνδεων. Αυτή τη μικρή διόρθωση θέλω να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ανθρώπινα τα λάθη, το διορθώσαμε. Λοιπόν, εδώ λίγη η δημόσια συνεδρίαση μαζί για σήμερα και θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να περάσουμε στην κεκλεισμένο των θυρών. Για να ακούσουμε τι γίνεται στους τριμερείς διαλόγους. Τα μέλη μπορούν να παραμείνουν, αλλά το κοινό ε, παρακαλείται να αποχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς μεγάλη τη λήψη. Στο καλό να πάτε.